τις κλινικές ε, δοκιμές φαρμάκων για χρήση σε ανθρώπους, για ανθρώπινη χρήση. Παρακαλώ πολύ. Wilmot. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης συζητητές για τη θαυμάσια στήριξη και συνεργασία. Μαζί καταφέραμε να επιτύχουμε πολλά για το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ και την Λιθανική Προεδρία για την τεράστια προσπάθεια που έκαναν για να καταλήξουμε σε συμβασμό έγκαιρα και την Κομισιόν που υπέβαλε καλή πρόταση και βοήθησε πάρα πολύ κατά τις συζητήσεις. Να ξεκινήσω με γιατί άρχισα να ασχολούμαι με αυτή την νομοθεσία πριν από τρία χρόνια. Πήγα σε ένα κέντρο για ε, παιδιά με όγκους στον εγκέφαλο. Είδα εκεί παιδιά στο Νότιγχαμ που είχαν σπάνιους καρκίνους και ένα νέο που λεγόταν Sam Μου είπαν ότι πολύ συχνά δεν υπήρχε θεραπεία για το πρόβλημά τους ε, έπρεπε να χρησιμοποιήσουν ε, φάρμακα που ε, έχουν δοκιμαστεί μόνο σε παιδιά και για πολλές σπάνιες ασθένειες δεν είναι δυνατόν να γίνουν κλινικές δοκιμές σε μια χώρα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολες και ακριβές αυτές οι δοκιμές. Αυτός ο νέος κανονισμός εναρμονίζει τους κανόνες σε όλη την Ένωση δημιουργεί μια διαδικασία για υποβολή αίτησης μέσω ε, πύλης και θα αλλάξει εντελώς την κατάσταση. Δυστυχώς ο Sam White ε, απεβίωσε πέρυσι το Σεπτέμβριο, αλλά συνεχίζεται η δουλειά που, με που μου ενέπνευσε και ελπίζω ότι αυτά που ε, επιτύχαμε θα βοηθήσει να βοηθήσουμε άλλους και θα αυξήσει την ε, βιωσιμότητα για αυτές τις σπάνιες ασθένειες. Αλλά όλες οι κλινικές δοκιμές πρέπει να βοηθούν σε καλύτερα φάρμακα. Μόνο μισές δημοσιεύονται αυτή τη στιγμή και πιο πιθανό είναι να δημοσιευθούν τα θετικά από τα αρνητικά αποτελέσματα. Οπότε δίνει μια μερική εικόνα για το πόσο αποτελεσματικά είναι κάποια φάρμακα και μπορεί να αναγκαίσει σε ε, άχρηστες ε, δοκιμές, επικάλυψη δηλαδή και ακόμη και επικίνδυνες δοκιμές να επαναλαμβάνονται. Όλες λοιπόν οι δοκιμές, θετικές, αρνητικές ή χωρίς αποτέλεσμα, θα πρέπει να δημοσιεύουν μια περίληψη των πορισμάτων τους σε ένα δημόσιο site. Και θα πρέπει μόλις, ξεκινάει, μόλις τελειώνει η δοκιμή να έχουμε τις εκθέσεις αυτές. Και βεβαίως δεν θα πρέπει να θεωρούνται εμπορικά εμπιστευτικές. Ελπίζω λοιπόν να υποστηρίξουμε την υπηρεσία για τα φάρμακα, το φορέα μας για τα φάρμακα στην προσπάθεια και χαιρόμεθα που στη διαφάνεια για τις κλινικές δοκιμές ε, παίζει πρωτοπόρο ρόλο η Ένωση. Αυτό είναι καλό για την ασφάλεια των φαρμάκων και για το κοινό. Αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κλινικές δοκιμές ε, διεξάγονται εδώ στην Ευρώπη, ούτως ώστε να υπάρχουν ευκαιρίες εδώ για νέες θεραπείες και να υποστηρίξουν χιλιάδες ειδικευμένε θέσεις εργασίας στην έρευνα. Ξέρουμε από το 2007 οι κλινικές δοκιμές ε, που γίνονται στην Ένωση μειώθηκαν κατά 25% και ελπίζω αυτό το νέο νομοθέτημα να βοηθήσει να μειωθεί η άχρηστη γραφειοκρατία και με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει ασφάλεια και σιγουριά και για τις εταιρείες και για τους πανεπιστημιακούς. Και επίσης θα προωθήσουμε τις ε, κλινικές δοκιμές μικρότερου κινδύνου. Αλλά καρδιά της νομοθεσίας είναι η προστασία των πελατών. Επιτροπές διοντολογίας πρέπει πάντα να συμμετέχουν στην αποτίμηση των κλινικών δοκιμών και να έχουν ε, την εξουσία να τις ε, διακόπτουν αν χρειάζεται. Επίσης έχουμε αναλυτικό κείμενο για την προστασία ευαλώτων τμήματων του πληθυσμού και πρέπει όλοι όσοι συμμετέχουν στις δοκιμές να λάβουν πλήρη ενημέρωση εκ των προτέρων. Φυσικά είναι συμβασμό αυτό που προτείνουμε. Σε ορισμένου τομεί θα ήθελα να έχω κάνει περισσότερα. Θα ήθελα να συμμετέχουν περισσότερο οι ασθενεί και βραχύτερου χρόνου έγκριση. Αλλά καταλαβαίνω ότι ορισμένα κρατημέλη είχαν ε, αντιρρήσει και νομίζω ότι ο συμβασμό που επιτύχαμε είναι εξαίρετο. Σα ευχαριστώ όλου που μα βοηθήσατε να φτάσουμε εδώ και ελπίζω συνολικά το Κοινοβούλιο να εγκρίνει σήμερα τον κανονισμό αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βίλμοντ. Το λόγο έχει ο Επίτροπος ε, κ. Μπόργ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Γουλμούτ και τους κοιόδης εισηγητές για τη σκληρή δουλειά που έκαναν και την αγαστή συνεργασία που είχαμε κατά την επεξεργασία αυτή τη τόσο σημαντική έκθεση. Θα συμφωνήσω με την εισηγήτρια. Θα προτιμούσα να είναι πιο φιλόδοξα τα συμπεράσματα, κυρίω για το χρονοδιάγραμμα, αλλά πιστεύω αυτό που έχουμε, διότι πρέπει να λειτουργούμε βάσει του εφικτού, είναι μια καλή συμβαστική λύση. Ε, απηχώντας αυτά που μόλι ακούσαμε από την εισηγήτρια, κάτι διάρκεια των διαπραγματεύσεων όλοι τονίσαμε ότι είναι προ όφελο των ασθενών το ότι ε, συμβεί στο μέλλον. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε ε, και όχι μόνο οι ευρωπαϊκέ φαρμακευτικέ εταιρείε θα υποφεληθούν από τη νέα νομοθεσία. Γιατί? Διότι είναι κλειδί οι κλινικέ δοκιμέ ε, για να κατασκευαστούν νέα φάρμακα, για να υπάρξουν νέε θεραπευτικέ αγωγέ που συμπεριλαμβάνουν ιστάμινα φάρμακα και συνήθω πολλέ φορέ βλέπουμε ότι για σοβαρά σοβαρές ε, παθήσεις, όπως μας είπε μόλις η συγγήτρια, οι κλινικές δοκιμές είναι μοναδική ευκαιρία που έχουν ε, οι ασθενείς. Ε, προωθώντα λοιπόν την έρευνα, εσωτερική έρευνα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις κλινικές δοκιμές μπορούμε να συμβάλλουμε σημαντικά και στην ανάπτυξη, αλλά και στη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Με το νέο νομοθέτημα επίσης αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο των τελευταίων ετών της μείωσης κατά 25% των ερευνών ενώ ε, έχουν έχει διπλασιαστεί το κόστος, οι απαιτούμενες δαπάνες για την ε, έρευνα. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι είναι επίγουσα η ανάγκη να δράσουμε, ούτω ώστε να παραμείνουν οι κλινικέ δοκιμέ, των οποίων ο αριθμό έχει μειωθεί κατά 90% τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα να προστατευτούν ε, όσοι υπάγονται σε αυτές τις κλινικές ε, δοκιμές. Ε, θα πρέπει λοιπόν να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των ασθενών, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσουμε τον αριθμό των κλινικών δοκιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτό το νομοθέτημα πιστεύω μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει η διαδικασία κατάθεσης αίτησης μέσα από ένα ενιαίο σημείο επαφής, μια ενιαία δικτυακή πύλη να διευκολυνθεί, να χρησιμοποιείται νέο έντυπο για να διευκολύνεται η επεξεργασία της αίτηση σε δεύτερο στάδιο για τις κλινικές δοκιμές, αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε επικάλυψη και ε, περίτη ε, καθυστέρηση. Στη συνέχεια έχουμε τη γνωστή αρχή ε, της ε, εγκεκριμένη ε, συμφωνίας για τη διαδικασία διοδότησης. Αυτό μας επιτρέπει, χειρώντα την ασφάλεια, να επιτρέψουμε στους σπόνσορες, κυρίως στις επιχειρήσεις και στους ακαδημαϊκούς κύκλους, να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία λοιπόν για την έγκριση για τη διαδικασία διοδότηση. Σε τρίτον, οι σπόνσορε δεν χρειάζεται χωριστά να καταθέτουν τι ίδιε πληροφορίε σε διαφορετικού εθνικού φορεί και σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Υπάρχει ομοιόμορφη διαδικασία. Επίση, αυξημένη διαφάνεια ε, για τι κλινικέ δοκιμέ, ακόμη και σε περιπτώσει όπου απορρίπτεται ή τροποποιείται ή και εγκρίνεται μία αίτηση. Και επιπροσθέτω, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, οι κλινικέ δοκιμέ που διεξάγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίε όμω ε, σχετίζονται με μια εφαρμογή κλινική δοκιμή που διεξάγεται εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η κλινική δοκιμή γίνεται εκτό όμω η αίτηση για την χορήγηση άδεια για ένα συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα κατατίθεται εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να συμμορφώνεται με κανονιστικέ απαιτήσει που θα είναι τουλάχιστον του ύψου αυτών που προβλέπονται στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλο ε, θα ε, είναι δυνατή η διεξαγωγή των ελέγχων τόσο σε κράτη-μέλη όσο και σε τρίτε χώρε, ούτω ώστε ε, να υπάρξει κατάλληλη εποπτεία και σωστή εφαρμογή των κανόνων για τι κλινικέ δοκιμέ. Εξαίρετοι μου κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και πάλι κλείνοντα να τονίσω πόσο σημαντική αυτή η νομοθεσία που θα ψηφιστεί στη συνέχεια, θα προωθήσει την κλινική έρευνα στην Ευρώπη και θα μα επιτρέψει να βρούμε λύσει για του ασθενεί για του οποίου προ το παρόν δεν υπάρχει διαθέσιμη θεραπευτική αγωγή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το λόγο έχει η πρόεδρος Αμαλία Σαρτόρη. Δεν παρίσταται η πρόεδρος Σαρτόρη, επομένω προχωρούμε. Το λόγο έχει η κυρία Αντωνία Παρβανόβα. Δεν είναι παρούσα. Bene, Επομένω, ο κύριος Φιλίπ Ζουβάν. Κύριε Πρόεδρε, ο κανονισμός για τις ε, ε, κλινικές δοκιμές μπορεί να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στην Ευρώπη για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί θα ε, είναι ίδια η διαδικασία διοδότησης για όλη την ενωσιακή επικράτεια. Δεύτερο σημείο είναι ότι οι διαδικασίες θα απλουστευθούν, ε, πράγμα που βεβαίως θα διευκολύνει ε, και ε, τα πανεπιστήμια κυρίως, αλλά και όλους όσους ασχολούνται με το ζήτημα αυτό και που βεβαίως θα υπάρχει πλέον ένας ενιαίος συνομιλητής και όχι πλειάδα συνομιλητών. Τρίτον, θα συντομεύσουν οι διαδικασίες, θα είναι πιο σύντομες και επομένως θα πλουστευτεί η ζωή των ερευνητών και των ακαδημαϊκών ερευνητών. Τέταρτον, θα δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα, όλα τα αποτελέσματα, ακόμα και τα αρνητικά αποτελέσματα, με επακόλουθη αύξηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δοκιμές αυτές. Τέλος, για πρώτη φορά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κίνδυνος ο οποίος προστίθεται στις ε, ε, δοκιμές αυτές θα λαμβάνεται υπόψη και όχι ο συνολικός κίνδυνος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, απλούστευση, επιτάχυνση ε, των διαδικασιών με ταυτόχρονη μείωση του κόστους και μεγαλύτερη προστασία για τους ασθενείς, μεγαλύτερη και γρηγορότερη εξέλιξη των διαδικασιών όσον αφορά τα αποτελέσματα και επομένως με μεγάλα πλεονεκτήματα για τον ε, ερευνητικό κόσμο αλλά και για τα ίδια τα σκευάσματα βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Έφτασε η κυρία Παρβανόβα και θα της δώσουμε το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Επίτροπε. Καταρχάς να συγχαρώ θερμά την για την εργασία της με θαυμάσιο τρόπο επέτυχε αποτελέσματα συλλογική εργασία για τα οποία μπορεί να είμαστε περήφανοι. Από πλευρά της ΣΥΜΚΟ και ως ε, σκιώδη για ένβη τη Άλντε θεωρώ ότι το νομοθέτημα αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα προς όλους τους τομείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με το μέλλον της έρευνας και ανάπτυξης. Η ασφάλεια, η διαφάνεια και η ελκυστικότητα ε, είναι τα βασικά στοιχεία που ε, προωθεί η πολιτική μου ομάδα και χαίρομαι που αντανακλώνται στο τελικό κείμενο. Πρέπει να προσελκύσουμε την έρευνα στην Ευρώπη ούτω ώστε οι πελάτες να υποφελούνται γρήγορα από την ανακαίνιση και πρέπει να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Θέλουμε διαφάνεια και αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση στοιχεία για την ε, δημόσια πολιτική και τις προτεραιότητες. Και τα επιτύχαμε όλα αυτά κατά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ Γκλένης για τη θαυμάσια αυτή συμφωνία που επέτυχε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έπαιξε αποφασιστικό ρόλο ούτως ώστε να βοηθήσουμε ε, τους ε, ασθενείς να ε, επωφεληθούν από καινοτόμα έρευνα. Ελπίζω να στηριχθεί και να εφαρμοστεί αυτό το νομοθέτημα που θα στηρίξουμε και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Παρμπάνοβα. Θα δώσω τώρα το λόγο ε, στον κύριο Ζουλ Παρνιό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα, Γκλένις, ε, για την εργασία που εκπώνησες ως εισηγήτρια, γιατί πλέον ε, ήταν επίγουσα η κατάσταση. Έπρεπε να υποβληθούν προτάσεις έτσι ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω μείωση ε, της υποβολής αιτήσεων για ε, ε, κλινικές δοκιμές οι οποίες τα τελευταία χρόνια είχαν πέσει κατά 25%. Διαπιστώσαμε επίσης ότι και το διοικητικό κόστος αλλά και οι πολύ μακρύ, μακρές προθεσμίες είχαν ανασταλτικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα. Επομένως είναι πολύ θετικό που το πλαίσιο για τις δοκιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται πιο πλέον πιο ευέλικτο. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχει ένα ε, βαρύ δημοσιον... Ε, διοικητικό και γραφειοκρατικό περίβλημα σε όλες αυτές τις ερευνητικές διαδικασίες και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η διαφάνεια και των ίδιων των δοκιμών αλλά και της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων, ε, σωστή πληροφόρηση και των ασθενών και αύξηση των προστατευτικών μέτρων που λαμβάνονται για τα πλέον ευάλωτα άτομα και βεβαίως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά ε, αποτελούν μεγάλη τιμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τα έχει περιλάβει σε αυτήν την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Παρνιό. Τον λόγο έχει η κυρία Όκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνεργαστήκαμε εδώ και πολλά χρόνια καλά και ήταν αρκετά σκληρές πραγματεύσεις. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για αυτή την καλή συνεργασία και ευχαριστώ γιατί υπάρχει διαφάνεια για την φαρμακοβιομηχανία και ελπίζω να υπάρχουν και αναγκαίες ε, προσπάθειες για να υπάρχουν οι επιτροπές ε, δεοντολογίες. Βεβαίως, πρέπει επίσης να μειωθεί και η τιμή των φαρμάκων που ε, εισάγονται στην αγορά. Δεν θα πω τώρα πώς θα πρέπει να λειτουργήσει αυτή η διαφάνεια, τα περιγράφει η έκθεση. Θέλω να διαπιστώσω ότι προέκυψε ότι οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, κυρίως οι αμερικανικές ε, φαρμακευτικές εταιρείες, θέλουν να καταργήσουν αυτόν τον κανονισμό, δεν θέλουν αυτούς τους κανόνες, γιατί δεν τις βολεύουν. Όχι όμως, εμείς θα επιμείνουμε γιατί στόχος μας είναι να μειώσουμε τις δαπάνες, να βοηθήσουμε τους ασθενείς και αυτά θα είναι και υπέρ των ασθενών στην τελευταία ανάλυση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Όουκεν. Μίλαν Καμπρόνκ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω τη δυνατότητα να παραστώ σημερινή συζήτηση που κλείνει ένα από τα πιο σημαντικά νομοθετικά πακέτα της ε, τωρινής θητείας. Ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με το Συμβούλιο, χάρη στην πρόταση του Κοινοβουλίου, ε, συντομεύεται σημαντικά η περίοδος που προβλέπεται για την ε, χορήγηση της έγκρισης. Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτές τις 60 ημέρες. Σας ελπίσουμε ότι δεν θα χρησιμοποιείται αυτή η ανώτατη προθεσμία κάθε φορά. Υπάρχει και η σιωπηρή διαδικασία φυσικά για τη χορήγηση έγκρισης όλα τα κράτη που θα μετάσχουν θα διαπιστώσουν ότι απλοποιείται η διαδικασία και έτσι έχουμε μια σημαντική ε, ευκαιρία να επιτύχουμε την επιστροφή της φαρμακευτικής έρευνας ε, στην Ευρώπη. Ε, θα, οι πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες στο νέο σύστημα θα είναι υποφελείς για όλα τα κράτη-μέλη αλλά και για τις φαρμακευτικές εταιρείες που θα έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα για τις αρχές λήψης αποφάσεων. Ευχαριστούμε κυρία Σούζα. Τώρα ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την Γκλένισε Βίλμοντ καθώς και τους κοιότητες εισηγητές διότι θεωρώ ότι η συνεργασία για αυτό το ζήτημα ήταν πάρα πολύ καλή και μας οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, κατά την γνώμη μου ε, και αξίζει την έγκριση από πλευρά του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα μια ερώτηση, ένα σχόλιο να κάνω πρώτα. Δεν ξέρω αν εκφράζομαι καλά, ε, ακόμη και στη γλώσσα μου. Λέμε στα πορτογαλικά Ε, ή μάλλον να στο πω αλλιώ, ε, είπατε ότι οι Ευρωπαίοι ασθενεί ε, θα υποφεληθούν από αυτή τη διαδικασία περισσότερο από ότι οι φαρμακευτικές εταιρείε. Ναι, αληθεύει αυτό, αλλά αυτό θα πρέπει να αποδοθεί στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η δική σα πρόταση επίτροπε, φαινόταν να έχει διατυπωθεί από την ίδια την φαρμακευτική βιομηχανία. Ε, χάρη στη δική μας δουλειά ε, κατοχυρώσαμε τη δουλειά των Επιτροπών Δεοντολογίας, ε, την διαφάνεια και την διαφύλαξη των δικαιωμάτων όλων όσων μετέχουν στη διαδικασία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι χάρη στην άσκηση της δικής μας μεικτής αρμοδιότητας που το καταφέραμε αυτό και όχι στη δική σας πρόταση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μόργαν. Μοργάντη, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ακόμα πολλές ασθένειες για τις οποίες δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία και επομένως καλωσορίζουμε τις δοκιμές και τα πειράματα. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ε, σε όλη αυτή την ιστορία ε, οι ασθενείς αυτοί που υποφέρουν και που προσβλέπουν σε κάποια ελπίδα, σε νέες μεθόδους, σε νέα φάρμακα τα οποία θα έχουν αποτέλεσμα. Αυτή είναι η προσδοκία, η ελπίδα που έχουν και στην Ιταλία ε, πάρα πολλές ε, οικογένειες οι οποίες ε, με τα βλαστοκύτταρα και με τις μεθόδους του καθηγητού Βανώνη προσπαθούν να δουν αποτελέσματα. Εγώ δεν είμαι ούτε ερευνητής ούτε επιστήμονας αλλά ήρθα σε επαφή με αυτές τις οικογένειες. Τις άκουσα προσεκτικά και έχω πλέον σαφείς απόψεις. Νομίζω ότι αυτές οι θεραπείες είναι η τελευταία τους ελπίδα και είναι κρίμα, είναι ντροπή που υπάρχουν ε, ε, γιατροί οι οποίοι δεν δέχονται, απορρίπτουν αυτές ε, τις ωστόσο καλά βασισμένες σε ιατρικές αρχές σε θεραπείες. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής 1,5 λεπτό είναι ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Σήμερα μπορούμε να είμαστε όντως ε, περήφανοι. Είναι πολύ συγκεκριμένη πρόοδος για τους ασθενείς στην Ένωση αυτό το οποίο καταφέραμε από κοινού. Πολλοί γιατροί, πολλοί ερευνητέ, πολλοί ασθενείς περίμεναν χρόνια. Τι περίμεναν, να μειώσουμε την γραφειοκρατία για τις διασυνοριακές κλινικές δοκιμές στην Ένωση. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει καλή έρευνα. Και αυτό ιδιαίτερα για τα ιδρύματα που είναι ανεξάρτητα από τη φαρμακοβιομηχανία, όπως ε, ο Οργανισμός για τη Βοήθεια στους Καρκινοπαθείς στην ε, Γερμανία, που θα ήθελε τις χρηματοδοτήσεις του να τις δαπανά όχι για γραφειοκρατία αλλά για έρευνα. Τα καταφέραμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κλένης Wilmot, καταφέραμε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Τα αρνητικά αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών δεν θα πρέπει να τα κρύβουμε. Και επίσης επιτύχαμε να υπάρχουν ισχυροί κανόνες δεοντολογίας. Αυτοί που είχαμε ήδη στην οδηγία. Διορθώσαμε την Κομισιόν και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Επίτροπο, Επίτροπο Μπόργ που ε, μας συνόδεσε αυτή την προσπάθεια. Η αρχική πρόταση δεν ήταν δική του. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τον Επίτροπο, ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν την Προεδρία, την εισηγήτρια, τους Κιώδης. Νομίζω ότι είναι καλό αποτέλεσμα και ελπίζω να υπάρξει ε, και ευρία πλειοψηφία κατά την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Ερχόμαστε στη διαδικασία προσέλκυσης της ε, προσοχής του Προέδρου και δίνω το λόγο στην συνάδελφο Κλάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι κλινικές δοκιμές είναι απαραίτητες για την έρευνα και για να υπάρχουν καλύτερα και νέα φάρμακα και θεραπείες. Με τις ε, δοκιμές μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι παρενέργειες των φαρμάκων πριν εισαχθούν στην αγορά. Οι δοκιμές είναι όμως και πολύ ευαίσθητο θέμα, γιατί τίθενται σημαντικά θέματα διοντολογίας, διαφάνειας και προστασία των ε, ευαλώτων ομάδων όπως είναι οι έγκοι, οι ανήλικοι και γι' αυτό είναι απαραίτητη αυτή η προσπάθεια κανονισμού. Οι κλινικές δοκιμές γίνονται σε δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη και η οδηγία είχε πολλές, ε, πολλά κενά και δεν εφαρμοζόταν από όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό χρειαζόταν εναρμόνιση. Ο κανονισμός οπωσδήποτε μειώνει και την γραφειοκρατία. Ο συμβασμός λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των ε, ενεχομένων. Χωρίς την έγκριση των επιτροπών διοντολογίας δεν θα μπορούν να γίνονται κλινικές δοκιμές και η διευκρίνηση του ρόλου αυτών των επιτροπών διοντολογίας είναι σημαντική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και τους την εισηγήτρια λοιπόν και του κοιόδης και ελπίζω αύριο να ε, ε, τύχει ευρεία αποδοχής. Ευχαριστώ ε, κυρία συνάδελφε. Κουρέα του Κάμπους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι λυπάμαι που δεν εγκρίθηκαν διατάξεις ε, χάρη στις οποίες θα ήταν δυνατές ε, και συνεργατικές ε, κλινικές δοκιμές που είναι απαραίτητες όμως για την αποτίμηση των νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Παρόλα αυτά υπήρξαν πολλά ρηξικέλευτα στοιχεία σε εναρμονισμένη διαδικασία αδειοδότηση σε διακρατικού χαρακτήρα για να αποφύγουμε την περιττή γραφειοκρατία, σύσταση ενιαίας δικτυακής πύλης όπου συγκεντρώνονται όλε τι πληροφορίε από όλε τις κλινικές δοκιμές, από όλου του εθνικούς φορείς ε, ταξινόμηση των κλινικών δοκιμών ανάλογα με το βαθμό παρέμβαση, ο ρόλο των εθνικών φορέων και επίση συγκεκριμένε απαιτήσει σε σχέση με τη δημοσίευση τη έκθεση τη κλινική δοκιμή. Οι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, βελτίωσαν σε μεγάλο βαθμό την αρχή πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την συνάδελφό μου Γκλένη Βίλμοντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στηρίζω αυτή, αυτό το νομοθέτημα, έστω και αν υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ε, ε υπολείπονται αποτελεί ένα καλό σημείο αναφοράς ε, αυτό το, αυτή η διαδικτυακή πύλη και νομίζω ότι είναι κάτι ε, πολύ θετικό έτσι ώστε να ξεπεραστούν ε, τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Το πνεύμα της εκθέσεως με βρίσκει σύμφωνο γιατί θα πρέπει οι ασθενείς, θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μπορούν να βρουν ανακούφιση σε καλά δοκιμασμένα συγκεκριμένα φάρμακα να έχουν δυνατότητα πρόσβαση στα φάρμακα αυτά. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί. Ε, δεν ε, ε, μπορώ να συμφωνήσω με την μία αναφορά των ζημιών που μπορούν ε, να προκύψουν ε, και βεβαίως με τον τρόπο αυτό θα μείνουν απ' έξω πολλές δοκιμές που μπορεί να είναι σωτήρες για την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ. Πατράου Νέβης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους σκιώτες εισηγητές για αυτή την έκθεση. Είναι εξαιρετική δουλειά που έκαναν. Ε, χάρη στη δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιφέραμε σημαντικότητα τη βελτιώσει στην αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ω προ τα πλεονεκτήματα τώρα τη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ταχύτητα ε, τη διαδικασία, ε, τη μείωση ε, του κόστου ε, και εν γέννη τη εγκαθίδρυση ε, νέων συνθήκων που προάγουν την επιστημονική έρευνα, έχουν υποθεί ήδη αρκετά κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Όμω, ταυτόχρονα θα πρέπει να τονίσουμε πώ υπήρξε μια μέλη στην οδηγία του 2001 για τα θέματα διεοντολογίας ε, και ε, χάθηκε αυτή η διάσταση στην αρχή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, αποκαταστάθηκε όμως η ισορροπία με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι τώρα αλλά στο μέλλον θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιτύχουμε πρόοδο στην επιστημονική και έρευνα, αλλά να μην ξεχνάμε τους κανόνες διοντολογίας που προστατεύουν τους όσους μετέχουν στις επιστημονικές κλινικές δοκιμές. Σας ευχαριστούμε. Και τελευταία στη διαδικασία προσέλιξης προσοχή, η κυρία Μπότσαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τα νέα φάρμακα, οι νέες ε, μέθοδοι θεραπείες μπορούν να σώσουν ζωές. Πριν από αυτό όμως ε, θα πρέπει να περάσουν από μια ε, διαδικασία, τη διαδικασία των κλινικών δοκιμών. Και αυτές οι κλινικές δοκιμές στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρουν, εμπίπτουν σε διαφορετικούς κανονισμούς, υπόκεινται μάλλον σε διαφορετικούς κανονισμούς. Ε, το ε, σύστημα των ε, θεραπείων θα αλλάξει. Η στάση των ασθενών αλλά και των γιατρών μέσα από καλύτερες κλινικές δοκιμές θα αλλάξει επίσης. Θα πρέπει βέβαια να προστατευθούν η ασφάλεια και τα δικαιώματα των ασθενειών. Υπάρχουν όρια τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν θα πρέπει να γίνονται γνωστές ε, βέβαια και οι δοκιμές οι οποίες έχουν αποτύχει, έτσι ώστε να μην χρηματοδοτούνται δοκιμές οι οποίες έχουν ήδη αποτύχει. Ωραία, Έληξη διαδικασία προσέλκυσης προσοχής και να δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Μπόρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους Κιώδης για την ε, δέσμευσή τους και την έντονη δουλειά που θα βοηθήσει την ε, ιατρική έρευνα στην Ευρώπη και θα διασφαλίσει όμως και υψηλή προστασία. Όταν μια πρόταση είναι καλή και μετά βελτιώνεται από το Κοινοβούλιο δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλή στην αρχή. Αυτή είναι η δημοκρατική διαδικασία. Μια καλή πρόταση βελτιώνεται. Για παράδειγμα. Και δεν ε, νύπτω τα σχήρα μου για την Κομισιόν συνολικά γιατί θα μπορούσα να πω ότι δεν ήμουν εδώ όταν έγινε η πρόταση αλλά όχι πρέπει να υπερασπιστώ συνολικά την Επιτροπή. Στην αρχική πρόταση για τις Επιτροπές Δοντολογίες, επειδή είναι κανονισμός, δεν ήθελε η Κομισιόν να επιβάλλει συγκεκριμένη δομή για όλα τα κράτη-μέλη για αυτές τις Επιτροπές, γιατί υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις. όταν κάποιοι ευρωβουλευτές και κάποιοι υπουργοί, πρέπει να πω, συζήτησαν το θέμα μαζί μου, τότε αμέσως συνέβαλα στην βελτίωση του κειμένου. Αναφέρθηκα στα θέματα διοντολογίας, γιατί βεβαίως εγώ ε, ως Επίτροπος ενδιαφέρομαι πολύ για να υπάρχει η καλύτερη διοντολογία. Λόγω λοιπόν της νομοθετικής διαδικασίας γίνονται βελτιώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αρχική πρόταση συνετάχθη από την φαρμακοβιομηχανία. Πολύ περίεργο είναι να λέγεται κάτι τέτοιο γιατί υπενθυμίζω κύριοι βουλευτές, η αρχική πρόταση είχε υποχρεωτική συμμετοχή των ασθενών στην αποτίμηση των ε, φαρμάκων. Ήταν η πρώτη φορά που ε, προτινόταν κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν η αρχική πρόταση και μετά νομίζω αφαιρέθηκε κατά τον τριμερή διάλογο από κάποια κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Και επίσης η αρχική πρόταση της Κομισιόν πρότεινε ε, δωρεάν ε, εθνικούς μηχανισμούς αποζημιώσεων. Αλλά ε, βεβαίως επειδή έπρεπε κάτι να επιτύχουμε χρειάστηκε να αποσύρουμε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Θέλω λοιπόν να υπερασπιστώ την αρχική πρόταση της Κομισιόν η οποία, σημειώνω, με ικανοποίηση βελτιώθηκε. Χαίρομαι λοιπόν που είμαι παρόν όταν καταλήγει η συζήτηση για αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω ότι θα διευκολύνει τις κλινικές δοκιμές στην Ευρώπη, όχι εκτός, και επίσης θα ωφελήσει την έρευνα, άρα και τους ασθενείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Μπόρτς. Και τώρα να δώσω και πάλι το λόγο στην εισηγήτρια συνάδελφο Wilmot. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους ομιλητές ε, που συνεισέφεραν σε αυτήν τη συζήτηση. Ε, και ε, όπως είπε προηγουμένως και ο Επίτροπος Μπόργκο, το κέντρο, το επίκεντρο της προσοχής μας είναι και πρέπει να είναι ε, ο ασθενής. Ε, θέλουμε να υπάρχει μικρότερη γραφειοκρατία, γι' αυτό ακριβώς δημιουργείται αυτή η ενιαία διαδικτυακή πύλη, έτσι ώστε ενώ διατηρούμε την ασφάλεια των ασθενών, κάνουμε πιο γρήγορη και πιο απλή τη διαδικασία. Αυτό είναι το σημαντικό σε τούτο νομοθέτημα. Μεγαλύτερη διαφάνεια Είπαμε ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών θα δημοσιεύονται ε, ακόμα και όταν είναι αρνητικά και όταν πρόκειται ε, για αποτυχία. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό για την υγεία και ε, θα αυξήσει οπωσδήποτε και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα πω δύο λόγια για τη στήριξη που είχα από όλους Ποτέ μέχρι τώρα δεν ε, είδα στο Κοινοβούλιο τόση συνεργασία και τόση καλή δουλειά. Στήριξη ε, της ε, εισηγήτριας, στήριξη από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο, αγαστή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών. Νομίζω ότι επιτύχαμε ένα πραγματικά καλό κείμενο, μια πραγματικά καλή ε, συμφωνία σε πνεύμα καλής συνεργασίας. Μακάρι όλα τα νομοθετήματα να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστώ κυρία Βίλματ. Λίγη συζήτηση, ψηφοφορία θα γίνει στις 6 ε, ώρα. Το επόμενο θέμα της μέρας διάταξης είναι η κοινή συζήτηση για τις ε, ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Με βάση την έκθεση της συναδέλφου Καστίγιο Βέρα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά και επίσης την έκθεση Herzog για τη μείωση